Ε, τώρα για την γνωμοδότηση του κυρίου Σταυρακάκη. Είμαι αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή ε, περιφερειακής ανάπτυξης και προσπαθώ να συμμετάσχω στο μέτρο δυνατού στις συνεδριάσεις της Επιτροπής και θα πω ε, εν γέννη για να μην πω σε λεπτομέρειες ότι αρχίζει η Επιτροπή να εξετάζει σοβαρά το θέμα των συνεργειών και της πιο αποτελεσματικής χρήσης των κονδυλίων. Αυτό δεν είναι νέο στοιχείο. Έχει προτείνει ήδη, ήδη τις νέες προσεγγίσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, πρώτον, η συμφωνία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κράτη θα συνάψουν δηλαδή συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποτελεσματικότητα ε, των ταμείων. Για τα έξι σημεία τίποτα ρίξει και έλευθο. Το ΕΚΤ ε, θα είναι μέρος της πολιτικής συνοχής, δεν θα ε, ε, λειτουργεί ξεχωριστά. Ίσως αυτό αντιτάσσεται στο γενικότερο στόχο. θέλω να σχολιάσω την πρόταση του κυρίου Σταυρακάκη να μπει και το γεωργικό ταμείο μέσα. Νομίζω ότι είναι λίγο προβληματικό αυτό δεδομένες της κατάστασης. Γνωρίζετε όλοι, τα γεωργικά κονδύλια έχουν διαφορετικά χρονοδιαγράμματα εκταμίευσης. Η συμφωνία ισχύει για 10 χρόνια, ενώ εμείς εδώ μιλάμε για 7 ετία. Πρότεινα προφορικά στον κύριο Σταυρακάκη γιατί θα υιοθετηθεί ε, τη η γνωμοδότηση το Φεβρουάριο, να σκεφτεί πώς ακριβώς μπορεί να υπάρχει συνέργεια με τον ε, πυλώνα 2 ε, στη Γεωργία, την ανάπτυξη της υπαίθρου δηλαδή. Από δημοσιονομικής πλευράς έχουμε τη δυνατότητα να δούμε αν δεν χρησιμοποιούνται ε, χρηστά τα κονδύλια. Το 70% δεν εκταμιεύτηκαν από πιστώσεις πληρωμών, δηλαδή το 2009. Τα κονδύλια πήγανε στο σχέδιο ανάκαμψης. Μετά το 2010 προσπάθησαν να τις ε, ξαναβρούν, ε, να ξαναβρούν αυτά τα πόσα που δεν εκταμιεύτηκαν. τώρα με το προπελισμό του 2010 του κυρίου Σούριαν, λέμε ότι πάλι τα παίρνουμε τα λεφτά από την αγροτική ανάπτυξη και τα πάμε στη συνοχή. Αυτή είναι η πρότασή μου και ελπίζω ότι θα πετύχουμε μεγαλύτερη συνέργεια ανάμεσα στο στα κονδύλια του δευτέρου πυλώνα της ε, Γεωργίας και το διαρθρωτικά ταμεία. Τα υπόλοιπα είναι φιλοσοφικά. Επιδιώκουμε περισσότερε συνέργειε. Σήμερα σε μια ε, συνεδρίαση τη Επιτροπή Ανάπτυξη των Περιφερειών είχαμε εκπροσώπου διαφόρων φορέων που μα εξήγησαν τα προβλήματα που υπάρχουν για τα διάφορα συστήματα διαχείρισης σε κάποιες χώρες ε, το ΕΚΤ και το ΕΤΠΕ την χάνουν διαφορετικής από τη δημοσιονομική πλευρά, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, θα πρέπει να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα. Πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια, δηλαδή. Και νομίζω ότι θα παραμείνουμε σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, να συντονίσουμε καλύτερα τα υπάρχοντα ταμεία και μελλοντικά, αν η ΓΑΜΑ κάνει πρόταση για πιο αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα στο δεύτερο πυλώνα της γεωργίας και τα διαρθρωτικά ταμεία Ίσως ε, μπει αυτό στην ημερήσια διάταξη, αλλά για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, εδώ αυτά είχα να πω. Ευχαριστούμε κυρία Κοντμανής. Ο συνάδελφός μας, το ξέρουμε ότι είναι απολύτως εμπειρογνώμονας αυτών των πολιτικών ε, και παρακολουθεί με θαυμαστό τρόπο τις ε, πιστώσεις και είναι σαφές και το βλέπουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη οικονομική θέση, κατάσταση γνώμη πολλών χωρών αντιμετωπίζουμε επιπλέον ε, πρόβλημα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των διαφορετικών ε, ταμείων. Ο συνάδελφος Βόν έχει ζητήσει το λόγο. Πολύ σύντομα. Πριν από λίγες μέρες είδαμε την ε, δημοσίευση της ε, πέμπτης έκθεσης ε, για το Ταμείο Συνοχής. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι οι περισσότερες από τις περιοφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι επιλέξιμες ε, για τα διευθυντικά ταμεία ε, και ενδεχομένως όντως μπορεί να υπάρχουν κάποιες διακοιμάνσεις όσον αφορά το ΑΕΠ και ότι επίσης το, το κοινωνικό ταμείο θα πρέπει να παραμείνει στην συνοχή. Όσον αφορά τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ όλων των των ταμείων και των διευθυντικών ταμείων νομίζω ότι είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε πάντως. Συμμερίζομαι την άποψη του κυρίου Γκουτμάνης ε, ότι δηλαδή δεν πρέπει να βάλουμε αυτή τη στιγμή την ανάπτυξη της υπαίθρου, το πρόγραμμα δράσης για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Ε, συμφωνώ με τον κύριο Κουτμάνης ότι δεν πρέπει να μπει αυτή τη στιγμή στα διευθυντικά ταμεία. Merci, mon cher collègue. Ευχαριστώ συνάδελφε. Άλλες παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κοντμάνης, έχετε να πείτε κάτι άλλο. Όχι. Όχι, ευχαριστώ. Ωραία λοιπόν. Είναι δύο οι εκθέσεις. Διαφορετικά ταμεία και ταμείο συνοχής. Η δεύτερη είναι πολύ πιο δύσκολη η έκθεση αυτή. Όπως είπε και ο κύριος Καρίγα, όλοι μας διαβάζουμε τους Financial Times. Η πρόταση αυτή του κυρίου Μικολάζεφ για την εφαρμογή των προγραμμάτων μέχρι το 2013 στα πλαίσια της ε, περιφερειακής πολιτικής. Εγώ προτείνω κάποιες αλλαγές που είναι καθαρά οικονομικού χαρακτήρα. Ένα, μπορούμε να εξασφαλίσουμε Καταρχήν βλέπουμε ότι η απορρόφηση είναι δύο φορέ χειρότερη από ό,τι στο παρελθόν. Δεν είναι θετικά νέα αυτά. Δυστυχώ για μερικά κράτη-μέλη μπορείτε να δείτε αυτή τη μεγάλη διαφορά στην ε, εκτέλεση των προγραμμάτων. Παραδείγματο χάρη για το κοινωνικό ταμείο πάνω από 57% των κρατών, 100 των κρατών μελών είναι κάτω από το μεσόωρο που είναι μόνο 19,9% και είμαστε στον πέμπτο χώρο. Για το Περιφερειακό Ταμείο και το Ταμείο συνοχή από κοινού 57% είναι κάτω από το μέσο όρο που είναι πάλι μόνο 19%. Το χειρότερο όμως είναι στο σημείο 3 των προτάσεών μου. Στο σημείο 4, συγγνώμη. Ο, η διαφορά μεταξύ καλών και κακών. Στον περιφερειακό τομέα δύο μισή φορές χειρότερος είναι ο ρυθμός απορρόφησης στο χειρότερο κράτος σε σχέση με το καλύτερο. Και τρεις φορές η διαφορά για το Ταμείο Συνοχής. Δυστυχώς, αν δείτε ποιες είναι οι διαφορές μέσα στο, στο χρόνο, κάποια κράτη-μέλη μπλοκάρουν απόλυτα, στομώνουν μέσα στους πρώτους μήνες του 2010 πρέπει να πω ότι δεν είχα προβλήματα συγχρηματοδότηση, γιατί βλέπουμε ότι τα χειρότερα αποτελέσματα είναι για τις χώρες που δεν έχουν μεγάλα ελλείμματα του προπολογισμού και μεγάλα χρέη. Σε τελική ανάλυση δεν μπορώ να πω τίποτα, το, δεν μπορώ να πω πολλά θετικά πράγματα. Η μόνη ελπίδα είναι ότι το 2011 και το 2012 θα υπάρξει μια βελτίωση. Αυτά που είπε και ο κύριος Επίτροπος ήταν θετικό. Είπε ότι το ποσοστό των σφαλμάτων μειώθηκε από 11% σε 3%. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι χάνουμε περισσότερο χρόνο. Το τρισταδιακό σύστημα για την πιστοποίηση, για την, ε, το λογιστικό έλεγχο και την έγκριση δεν επιτρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Αλλά το σύστημα αυτό έχει λιγότερα λάθη. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα εγώ να πω είναι ότι θα ήταν καλύτερο να δείξουμε στην Γενική Διεύθυνση Περιφερειακών Θεμάτων της Κομισιόν ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των χωρών και πρέπει να βελτιωθούν τα πράγματα το 2011 και ίσως ο διορθωτικός προϋπολογισμός του 2010 αν τον εγκρίνουμε, θα βελτιώσει την κατάσταση μέχρι τις 91 Δεκεμβρίου του Ενεστώτος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι. Για το Ταμείο Συνοχής έχουμε κάπως διαφορετική κατάσταση. Είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι για τα διαφορετικά ταμεία και αντίθετα από ό,τι θα μπορούσε κανείς να πιστέψει δεν είναι οι πιο ζωρισμένες χώρες από έποψη προϋπολογισμού αυτές οι οποίες έχουν τους χειρότερου βαθμούς σε ό,τι αφορά την απορρόφηση των κονδυλίων. Πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση. Δεν βλέπω να θέλει κανεί το λόγο. Θέλω ευχαριστήσω τον κύριο Γκοντμανή. Σα υπενθυμίσω για τι δύο αυτέ εκθέσει που είναι εκθέσει για γνωμοδότηση προ την Περιφερειακή Επιτροπή στι 17 Δεκεμβρίου στι 10 το πρωί εκπνέει η προθεσμία για τροπολογίε στην Επιτροπή μας. Θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση του κ. Γκότμανής στις 27 Ιανουαρίου και την επαύριο θα λάβει χώρα η ψηφοφορία στην Περιφερική Επιτροπή και το Μάρτιο Θεού θέλοντος θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης σήμερα το απόγευμα γιατί θα επανέλθουμε αύριο σε 9 για τα άλλα σημεία. Η ε, γνωμοδότηση του κυρίου Γκουαλτιέρη και της κυρίας Νέινσκι για την ετήσια έκθεση σε σχέση με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια και ΠΑ 2009. Κύριε Γουαλτιέρη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η γνωμοδότηση ε, η οποία φέρει την υπογραφή μου μεν αλλά έχει εκπονηθεί έχει εκπονηθεί με την ε, εισηγήτρια κυρία, συνεισηγήτρια κυρία ε, Νίνσκι αναφέρεται στα σημεία αυτά του προπολογισμού τα οποία περισσότερο σχετίζονται με την έκθεση του Κοινοβουλίου ε, για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Βεβαίως επικεντρωνόμαστε περισσότερο στις σημαντικές εξελίξει οι οποίες έχουν λάβει χώρα σε αυτά τα πλαίσια υπό το φως των συμφωνιών της ε, Μαδρίτη και την απόφαση δημιουργίας ε, της Ευρωπαϊκής Μονάδας Εξωτερικής Δράσης. Υπογραμμίζεται βεβαίως η σημασία της συμφωνίας που επέτρεψε την ταυτοποίηση κάποιων ειδικών ε, γραμμών όσον αφορά τις εκπομπές και βεβαίως τις τρεις μεγαλύτερες αποστολές οι οποίες ε, οδηγούν προς την ε, ε, διαφάνεια την οποία θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όσον αφορά όμως πλέον και τις μικρότερες σημασίες αποστολές. Ένα άλλο σημείο το οποίο θίγει η έκθεση, η γνωμοδότηση μάλλον, αφορά το θέμα το, της πληροφόρησης του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις ε, δαπάνες του στρατιωτικού σκέλους ε, της ε, ΚΕΠΑ. Εμείς θεωρούμε ότι σαν, σαν πολιτικό όργανο του Ευρωπαϊκού... της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοβούλιο, θα πρέπει να έχει και οικονομικό στοιχεία όσον αφορά ε, τις ε, ε, δαπάνες έστω και αν αυτές οι δαπάνες τελικά εμπίπτουν στους εθνικούς προϋπολογισμούς γιατί μην ξεχνάμε ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχει και στον, στη χρηματοδότηση του πολιτικού σκέλους της ΚΕΠΑ και επομένως θα πρέπει να έχει την διοικητική διαχείριση όλων των προϋπολογισμών και για την ΚΕΠΑ και για το στρατιωτικό σκέλος. Επομένως, ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά το συνολικό κόστος των στρατιωτικών αποστολών μια και συγχρηματοδοτεί τις αποστολές αυτές σαν ένας εκ των βραχιών του προϋπολογισμού. Αυτά είναι τα βασικότερα στοιχεία της γνωμοδότησης. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα πιο εξειδικευμένα τα οποία ας πούμε αφορούν το ρόλο των ειδικών εκπροσώπων. Τη στιγμή που ε, αυτοί ε, τα τίθενται εκτός ε, της ΚΕΠΑ και επίσης υπάρχει και ένα άλλο γενικότερο σημείο το οποίο αφορά την αντίληψη της ΚΕΠΑ έξω από τον προϋπολογισμό και είμαστε εδώ στο σύνολο των ε, πολιτικών που σχετίζονται με την ΚΕΠΑ έστω και αν, ε, δηλαδή που ε, συνορίζουν ε, την ε, ΚΕΠΑ χωρίς όμως να εμπίπτουν ακριβώς στον προϋπολογισμό ΚΕΠΑ. Οι συμφωνίες της, Μαδρίτη, της Μαδρίτης καθώς επίσης και το έγγραφο σχετικά με τον υπολογισμό των δαπανών των αποστολών πιστεύουμε ότι θα οδηγήσουν σε πιο αποτελεσματική σχέση με, τις, με τα σκέλη του προϋπολογισμού, της βραχίωνος του προϋπολογισμού και βεβαίως θα μας οδηγήσουν και σε πιο αποτελεσματική ΚΕΠΑ. Ευχαριστώ. Υπάρχει και ένας άλλος από την παλιά φρουρά, ο Ζουάν Κολόν. Χειροκροτήστε τον. Ο Ζουάν Κολόν ήταν ο συντονιστής της Σοσιαλιστικής Ομάδος πριν από πολλά χρόνια όταν ήμουνα εγώ Σιδονία, δηλαδή ήμουνα εισηγητής του προπολογισμού. Τότε που, που με τον, να πει απόρριψη του προπολογισμού πετύχαμε πρόοδο στα δημοσιονομικέ στις δημοσιονομικές προοπτικές. Ο Ζουάν μας λείπει πάρα πολύ, αλλά έγινε διαμέσως πρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου της Καταλωνίας. Νομίζω ότι λείπει και από το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Καταλωνίας τώρα αυτή τη στιγμή. Καλώς ήρθε Ζουάν, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε βλέπουμε. Δεύτερη εισηγήτρια η Αντέσνια Νιένσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λίγα φωνή μονάχα έχω να προσθέσω σε αυτά που λέει ο συναδελφός μου κύριος Γκουαλτιέρη. Απλώς θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε, στον κύριο λόγο για τον οποίο το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να υιοθετήσει τη νέα ονοματολογία που προτείνει η Κομισιόν. Διότι οι περισσότερες μεταφορές πιστώσεων που συνδέονται με πιστέσεις, πιστώσεις συγγνώμη, πληρωμών και οι οποίες δεν έχουν πολιτική κρυά χρειάζονται οι πιστώσεις αυτές μια ταχεία εκτέλεση και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι μια ιδιαίτερα πρόσφορη πρόταση διότι με τον τρόπο αυτό εγγυάται την διαφάνεια κατά τη διάρκεια της ε, Χρηματοδότηση των διαφόρων αποστολών της ΚΕΠΑ, διατηρώντας όμως και τον έλεγχο του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια αυτών των αποστολών. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα άλλο τομέα, ότι η επιρροή αυτής της υπηρεσίας ξεπερνάει το άρθρο το οποίο αναφέρεται, το κεφάλαιο 1903 του προϋπολογισμού και σας δίνω σαν παράδειγμα το μέσο ε, σταθερότητος ή την ειδική, τον ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης αυτές οι τροπολογίες έχουν βοηθήσει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερος έλεγχος από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, Δεν θέλει κανείς το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω τους δύο συναδέλφους μας. Οίκοθε εννοείται ότι του χρόνου η έκθεση αυτή θα είναι πολύ πιο σημαντική και θα έχει μεγαλύτερη εμβέλεια. Το γεγονός ότι είμαστε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών δεν μας επιτρέπει να συμμετάσχουμε σε ένα σημαντικό γεγονός που είναι η γιορτή της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και οποία λαμβάνει χώρα σήμερα πολύ κοντά από εδώ στις Βρυξέλλες και θα ακολουθηθεί από ένα μεγάλο σημαντικό λόγο της κυρίας Άστον. Διότι 1η Δεκεμβρίου μετά από ένα χρόνο από την θέση σε εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας σύμφωνα με τους πολιτικούς στόχους που είχαμε όλοι στην καρδιά μας είναι fully fledged η δημιουργία αυτής της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και λειτουργεί. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους συναδέλφους, την κυρία και τον κύριο Γκουλτιέρη και την Ίγκε βέβαια. Η Ίγκε εμπόδισε τα πράγματα λίγα, τα καθυστέρησε, οι άλλοι προσπαθήσαν να επιταχύνουν την πολιτική συμφωνία στον τομέα αυτό, όπως γίνεται πάντα. Και αυτό αφορά και το νομοθετικό πακέτο. Φτάσαμε λοιπόν σε μια καλή λύση του χρόνου όμως αγαπητοί συνάδελφοι. Πιστεύω θα είναι διαφορετική η εκθεσή σας καταδεικνύων ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εξωτερική της προβολή έχει αλλάξει διάσταση. Έγινε πραγματικός ηθοποιός. Και μετά από την διάσκεψη κορφής του ΝΑΤΟ με παρουσία κρατών και κυβερνήσεων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης είπα, αντί να μείνει μόνο δύο ώρες μένει δύο μέρες για να ανταλλάξει απόψη με τον κύριο Φαν την κυρία Άστον και τον πρόεδρο Μπαρόσο. Ευχαριστώ λοιπόν. Εξαντλήσαμε την ημερήσια διάταξη. Να σας υπενθυμίσω την υποθεσμία κατάθεση τροπολογιών για την έκθεση αυτή 7 Δεκεμβρίου το μεσημέρι. 27 Ιανουαρίου θα εγκρίνουμε την τροποποιημένη έκθεση. Στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα εγκριθεί την 1η Φεβρουαρίου και το Μάρτιο μπορεί να γίνει ψηφοφορία στην Ολομέλεια και για τον προϋπολογισμό μας 2010, 2011 καλύτερα, το σχέδιο του προπολογισμού 2011 που ελπίζουμε να κρίνουμε μέσα στο 2010 έχει προθεσμία κατάσταση των προλογιών για τη νέα πρόθεση κομισιών στις 3 Δεκεμβρίου σε μεθαύριο λοιπόν το μεσημέρι. Ωραία, τέλος της συνεδρίασης, αλλά θέλω να μείνουν εδώ οι συγητές, οι συντονιστές. Και ευχαριστώ και την νομική υπηρεσία για την παρουσία της και κρατώ και του μέχρι στις 6.30. Πέρασε.